Να σας ενημερώσω ότι τα πρακτικά για το κείμενα τα οποία εγκρίθηκαν στις 24 και 25 Φεβρουαρίου είναι διαθέσιμα. Ε, υπάρχουν σχόλια από πλευράς ε, συναδέλφων. Αν όχι,